μέρες και να περιμένουν επιμέρες για να πάρουν λίγα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Τικάου, για ένα λεπτό.